Καλησπέρα σας. Έχουμε μια σειρά ερωτήσεων στην ημερήσια διάταξη προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα θα ακούσουμε τις ερωτήσεις από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Μάνφρετ Βέιντε, για ένα λεπτό από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, συνάδελφοι. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, υιοθέτησε μια νέα συμφωνία SWIFT και υπήρξε μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ αυτού. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα γνωρίζει ότι πολλοί πολίτες ανησυχούν για το θέμα των δεδομένων και της προστασίας των δεδομένων. Τι μέσα ελέγχου και εξισορρόπησης υπάρχουν ε, στα πλαίσια αυτής της ε, σημαντικής ε, συμφωνίας. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι ομόφωνα εγκρίθηκε αναθεωρημένη αυτή συμφωνία σήμερα από την Κομισιόν σε πλήρη συμμόρφωση με τις διασφαλίσεις για την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων με τις αρχές της αναλογικότητας και σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Η συμφωνία όπως έχει αυτή τη στιγμή σέβεται όλες τις αρχές ε, της Χάρτας των Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων και παρέχει διασφαλή όσον αφορά την ε, επεξεργασία των δεδομένων από τον πάροχο, επίσης διαθεσιμότητα των δεδομένων για αυτούς που ζητούν να χρησιμοποιήσουν ένδικα μέσα. Ε, υπάρχει λοιπόν ε, πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αυτό ε, σύμφωνα και με το ψήφισμα που εγκρίθηκε πέρυσι το Μάρτιο για την διάμεση συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούλς, α, όχι. Ο κύριος Βέμπερ, μια συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε, μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Σχετικά με το περιεχόμενο της συμφωνίας, ε, είπατε μερικά πράγματα. Ε, ποιε είναι οι συνέπειε και οι επιπτώσει αυτή τη συμφωνία για τι διατλατικέ σχέσει. Έχουμε κάποια εκκρεμή ζητήματα με, την, ε, με τις ΗΠΑ. Τι ρόλο θα παίξει αυτή η συμφωνία. Ναι, όντω είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορώ να σα πω ότι οι Αμερικανοί θεωρούν, αν όχι την πρώτη προτεραιότητα, μία από τι μεγάλε προτεραιότητε των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κρίσιμη η συμφωνία αυτή για τις σχέσει μα με τι ΗΠΑ. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 ε, σημαντικές συμφωνίες, ε, δεν, ε, σημαντικές, σημαντικές πληροφορίες δεν ήταν διαθέσιμες και αυτό δημιουργούσε προβλήματα στις διμερείς μας σχέσεις. Και Ακριβώς είχαμε υπόψη μας τις διατλαντικές σχέσεις όταν ε, υπογράφαμε αυτή τη συμφωνία. Οι διατλαντικές βεβαίως ε, σχέσεις μας είναι πάρα πολύ σημαντικές, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα παραμείνουμε πιστοί στις αρχές μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων. Το γεγονός πάντως είναι ότι τώρα έχουμε ε, καταλήξει σε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά και από ευρύτερη πολιτική σκοπιά πιστεύω ότι θα είναι σημαντική ότι ήταν σημαντικό ε, το ότι καταλήξαμε σε μια συμφωνία με τους Αμερικανούς εταίρους μας για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι συμπληρωματικές ερωτήσεις και απαντήσεις θα είναι μόνο 30 ε, δευτερόλεπτα. Δυστυχώς αυτός είναι ο κανόνας μας και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, ο κύριος Σούλτς. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεχίζοντας τις ερωτήσεις του συναδέφου Μάνφρεντ Βέμπερ στην παρέμβασή του. Η Επίτροπος Μάλμστρομ ενημέρωσε το Σώμα των Επιτρόπων ότι σε σχέση με το πώς έχουν οι διαπραγματεύσεις σήμερα υπάρχουν μεγάλες επιφυλάξεις από πλευράς του Σώματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτά που σήμερα απεφάσισε σίγουρα δεν είναι αυτά που το Ευρωκοινοβούλιο θα επιθυμούσε για ε, να σημειωθούν επαρκής πρόοδοι. Έχετε συνειδητοποιήσει κύριε Πρόεδρε ότι σήμερα εγκρίνατε κάτι που αν έτσι εφαρμοστεί και ακολουθηθεί θα οδηγήσει στο ότι απασχολούμενοι σε μια ιδιωτική επιχείρηση στην εταιρεία SWIFT θα έχουν περισσότερες ελεγκτικές αρμοδιότητες από ό,τι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μάλμστρομ σας ενημέρωσε για αυτά τα πράγματα. Αν ναι, πώς μπορέσατε και αποφασίσατε κάτι τέτοιο. Αν όχι, τότε γιατί δεν σας ενημέρωσε και δεν πληροφορηθήκατε από την κυρία Μάλμστρομ. Ευχαριστώ. Βεβαίω Βεβαίως μας ενημερώνει συνεχώς η συνάδελφος για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και σήμερα ακόμα ε, η Επίτροπος μας ε, πληροφόρησε το, την έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων. Επίσης μας είπε ότι είχε ε, πολύ έντονο διάλογο με πολλούς από εσά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρχαν ανησυχίε εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά σα κρατούσε συνεχώ ενήμερου για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Η Κομισιόν έχει ε, εκπληρώσει το ρόλο τη να διαξαγάγει τι διαπραγματεύσει. Ε, τώρα, ο δικό σα ρόλο είναι να εγκρίνετε ή όχι αυτή τη συμφωνία. Σα ε, παροτρύνω θερμά να ε, υπερψηφίσετε, γιατί η συμφωνία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Εξασφαλίζεται η προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων και η προστασία των δεδομένων, αλλά ε, ε, υπάρχει και θέμα ασφάλειας. Ε, πιστεύω ότι ε, έχουν γίνει πλήρω σεβαστά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα ο ρόλος σας είναι να εγκρίνετε ή μη την συμφωνία. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, γι' αυτό. Αλλά δεν ήταν η απάντηση στην ερώτησή μου. Γι' αυτό θα ξαναπροσπαθήσω πιο εξειδικευμένα να ρωτήσω και παρακαλώ να απαντήσετε πιο εξειδικευμένα. Η κυρία Μάλμστρομ στη συζήτηση που διεξήχθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τη λήψη απόφαση του Συλλογικού Σώματο των Επιτρόπων, σα ενημέρωσε, σα είπε ότι με το κείμενο το οποίο ω συμφωνία υποβάλλεται εγκυμονείται ο κίνδυνος να καταψηφίσει η Ευρωβουλή αυτή τη συμφωνία ή η κυρία Μάντσορ σας είπε με αυτό το κείμενο θα υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία στην Ευρωβουλή. Επαναλαμβάνω με κάθε ακρίβεια. Η κυρία Μάντσορ σας είπε ότι θα επιτευχθεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία ή σας είπε με αυτό το κείμενο δεν διασφαλίζεται κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα ήμουν ευγνώμων αν απαντούσατε εξειδικευμένα. Ευχαριστώ. Ε, η Επίτροπος Μάμστρομ δεν μπορεί να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο. Όχι, η ερώτησή σας ήταν αν η κυρία Μάμστρομ μου είπε ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και η αντίδραση του Κοινοβουλίου, αν θα ψηφίσει ναι ή όχι το Κοινοβούλιο. Ελπίζει φυσικά ότι θα ψηφίσετε υπέρ, διαφορετικά δεν θα είχε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις εκ μέρους της Κομισιόν. Πριν από την αρνητική ψήφο του Κοινοβουλίου, πριν από μερικούς μήνες, κάναμε μια πολύ ε, σημαντική μια πολύ σοβαρή συζήτηση στην Κομισιόν. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά και η ίδια η επίτροπο προσωπικά έχει πλήρη επίγνωση του θέματο, γιατί έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και ξέρει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με αυτή τη συμφωνία αλλά φυσικά τώρα δεν μπορούμε εμεί να προβλέψουμε και να προδικάσουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα τη ψήφου στο Κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να μου το έχει πει. Μου είπε όμω ότι ε, έχουν γίνει διαβουλεύσει με το γενοβούλιο και δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σχετικά με το πότε θα γίνει η ψηφοφορία για την προτινόμενη αυτή συμφωνία. Αυτό μόνο μπορώ να σας πω ε, σχετικά με τις πληροφορίε που μου έδωσε η αρμόδια επίτροπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς μικρόφωνο οι ομιλητέ. Μήπως ε, θα προσκρούστε σε ένα όχι άλλη μια φορά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Πρόεδρος Βέρχοφστατ. Όχι, όχι, δεν θα θέσω ερώτηση για το SWIFT, θα το συζητήσουμε αργότερα. Αλλά χτες η κυρία Έρκελ Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή είχαν σύνοδο συνάντηση κορυφή και αποφάσισαν μια προσέγγιση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση και όχι στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι μια απόφαση που είναι πολύ χρήσιμη και συναφή, γιατί για μένα δεν είναι ένα θέμα της Ευρωζώνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη ευρώ. Χρειαζόμαστε και στα δύο ευρωπαϊκή διακυβέρνηση και στην Ευρωζώνη ακόμα πιο εντατική διακυβέρνηση εφόσον έχουμε το ενιαίο νόμισμα. Η ερώτησή μου κύριε Πρόεδρε είναι ποια είναι η άποψή σας. Συμφωνείτε μαζί μας ότι χρειάζεται οικονομική διακυβέρνηση και στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, σχετικά με αυτόν που θα καθοδηγεί αυτήν την ε, οικονομική διακυβέρνηση. Είμαστε τη γνώμη ότι η Κομισιόν πρέπει να το κάνει. Ένα συμβούλιο που συνεδριάζει τέσσερι φορέ το χρόνο δεν μπορεί να ασχοληθεί με τη διακυβέρνηση με όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε. Η Κομισιόν πρέπει να είναι στη θέση του οδηγού. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής σχετικά με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, κύριε Βερχοφστάντ, όσον αφορά στις αρμοδιότητες οι οποίες ήδη, τις οποίες έχει ένωση, η Κομισιόν είναι η οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης. Είναι η μόνη απάντηση η οποία συνάδει με τις συνθήκες σχετικά με το εμπόριο, τον ανταγωνισμό, ε, ένα σημαντικό μέρος ε, της ε, δημοσιονομικής επιτήρησης και εποπτείας. Πρέπει πολύ συχνά να το υπενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις μας που δεν διάβασαν αρκετά καλά με αρκετή προσοχή τις συνθήκες. Βεβαίως η Κομισιό μόνη της δεν μπορεί να επιτελέσει αυτό το έργο. Πρέπει να συμφωνεί με το Συμβούλιο και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που δίνει την γενική κατεύθυνση στις εργασίες της Ένωσης και συμφωνώ επίσης με την πρώτη σας δήλωση, όντως έχουμε την απάντηση για τη ζώνη ευρώ και για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο άρθρο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπει δυνατότητες ευρύτερες να έχουμε προτάσεις για την Ευρωζώνη διότι υπάρχουν, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην Ευρωζώνη και επιπλέον ε, να έχουμε ε, περισσότερα ε, μέτρα για αυτούς που έχουν το ενιαίο νόμισμα, αλλά επίσης και διακυβέρνηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να την ενισχύσουμε, αλλά πάντοτε τηρώντας το πνεύμα της συνθήκης και την κοινοτική μέθοδο. Πρόσθετη ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως. Ε, το πρώτο τεστ, η πρώτη δοκιμασία θα είναι την Πέμπτη όταν ληφθεί και η απόφαση για την Ευρώπη 2020 και ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι στην Ευρώπη 2020 ε, δεν είναι το Συμβούλιο που θα κάνει το monitoring, την επιτήρηση θα το κάνει η Κομισιόν διότι ποτέ δεν έχω δει αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που αρχίζουν να ε, τιμωρούνται αμοιβαία, να αλληλοκατηγορούνται μεταξύ των ομοτήμων. Αυτό δεν γίνεται και νομίζω ότι η Κομισιόν πρέπει να υπερασπιστεί τις θέσεις εδώ στην Ευρώπη 2020 ε, και ε, στην ομάδα εργασίας ε, που δημιουργεί ο κ. Φαντρομπέι. Κύριε Βερχοφστάντη, ήσασταν μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, γνωρίζετε καλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ένας θεσμός πάρα, πάρα πολύ σημαντικός, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε micromanagement ε, την οικονομική πολιτική διαμέσου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήταν μοιραίο σφάλμα, ε, βασικό θεμελιώδες σφάλμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο βεβαίως δίνει την όθηση, την καθοδήγηση βάση του άρθρου 16 και μετά τα άλλα όργανα, η Κομισιό με τις αρμοδιότητές της και το Συμβούλιο με τις δικές του πρέπει να εξακριβώσουν, να ελέγξουν την εκτέλεση των πολιτικών και βεβαίω η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να παίξει πλήρω το ρόλο τη σχετικά με την επιτήρηση τη διαδικασία 2020. Περιμένουμε την υποστήριξη των κρατών μελών για αυτή την στρατηγική. Με ενθαρρύνουν οι συζητήσει μέχρι τώρα και περιμένω και τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι θέσει του Κοινοβουλίου μα υποστηρίζουν πολύ, αλλά η Κομισιό είναι έτοιμη να παίξει πλήρω το ρόλο της. Θα ήθελα κλείνοντας κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω ειλικρινά για την σαφή θέση που οι τέσσερις βασικές ομάδες του Κοινοβουλίου εξέφρασαν στην συνέντευξη τύπου για την τήρηση του πνεύματος συνθήκης της Λισαβόνας. Η κυρία Ρεμπέκα Χάμς παρακαλώ. <clears throat> Αλλαγή θέματος, κόλπος του Μεξικού. Water, Deep Water Horizon. Είναι μια έννοια αυτή αυτής της πλατφόρμας και αυτού του ατυχήματος που τους ανθρώπους παγκόσμια τους ε, δείχνει ποια είναι τα όρια της ανάπτυξης και της πρόοδου και της ανάπτυξης και της διασπάθησης πετρελαϊκών πόρων και της αντιπαράθεσης ανθρώπων και τεχνολογίας. Θα ήθελα να ξέρω ως προς αυτό κύριε Παμπαρόζο ποιες είναι οι απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρόνοια πρέπει να λαμβάνεται προληπτικές δράσεις εκεί που είναι αρμόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνεται πρόνοια για τις σχεδιαζόμενες αυτές ενέργειες στη Βόρεια Θάλασσα με παρόμοιες πλατφόρμες να απαγορευτούν οι δράσεις. Τώρα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε αν πραγματικά πιστεύετε ότι οι ρυθμίσεις, οι διατάξεις που έχουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου μας προστατεύουν αυτές οι διατάξεις από επανάληψη τέτοιων καταστροφών σε θέματα που είμαστε αρμόδιοι. Ευχαριστώ. Στο πολύ για την ερώτησή σας. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους ε, μια και βρίσκεται υπό εξέλιξη η έρευνα. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια ήταν τα αίτια, αν ήταν φυσικά αίτια ή ήταν λήψεις ε, και κάποια κενά που υπήρχαν από πλευράς τεχνολογίας και βιομηχανίας. Γι' αυτό για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά την Ευρώπη αυτό δεν έχει κλείσει. Ενώ μπορούν να γίνονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στον κόλπο του ε, Μεξικού πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου είδους ε, ε, περιπτώσεις. Παρότι είναι ρηχότερα τα οπιθμένα της θάλασσας, στη Βόρεια Θάλασσα. Έχει ήδη συγκαλέσει τον Μάιο και συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες σε αυτά τα ύδατα για να έχουμε μια σαφή απεικόνηση τι συμβαίνει στην Ευρώπη και να έχουμε σαφεί διασφαλίσει για τα επίπεδα ασφάλεια. Εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη και την άμεση αντίδραση για να προστατευτούν όλοι οι, Ευρωπαϊκοί, οι Ευρωπαίοι πολίτε και το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Επερώτηση παρακαλώ εσείς, παρακαλώ. Η ε, κυρία Χάμ, θα σας παρακαλούσα να μου πείτε αν, σημαίνει ότι η οδηγία περί για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τέτοιου είδους πετρελαϊκή ρήπανση είναι επαρκής. Ή αν πιστεύετε ότι τα χαμηλά επίπεδα, ανώτατα επίπεδα είναι εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε δεδομένης αυτής της, καταστροφή της καταστροφής στον κόλπο. Και θα ήθελα να ξέρω αν συζητείτε εσείς ώστε τεχνική έλεγχη για τέτοιου είδους πλατφόρμες πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν. Και αυτό για το πρώτο θεματικό πλέγμα με οδηγεί πάλι σε αυτό. Πιστεύετε ότι το περιβάλλον και οι κλιματικές προϋποθέσεις στην Αρκτική είναι αρκετά φιλικές προς το περιβάλλον και προς τους ανθρώπους ώστε για την άντληση πετρελαίου υποθαλάσσια να συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι το ίδιο βάθος εκεί όπως στον κόλπο του Μεξικού αλλά οι συνθήκες είναι πάρα πολύ σκληρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα Υπάρχουν ε, ε, πρότυπα και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υπεράκτη άντληση, τον, την ασφάλεια του εξοπλισμού, του προσωπικού, την πρόληψη ατυχημάτων και την ετοιμότητα. Επιπλέον τα κράτη-μέλη έχουν ε, και δικιά τους ε, ε, ευρύτατη εθνική νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Δεύτερον, έχουμε ένα σύστημα άμεσης ανταπόκρισης που έχει σαν σκοπό να αποτραπούν τέτοιες καταστροφές από διαρροές κλπ. Αυτό το σύστημα το ε, διευθύνει ο Ευρωπαϊκός Αναφυλιακός Οργανισμός. Τρίτον, υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, προστασίας που μπορεί να απαντήσει σε κάθε μια τέτοια επίγουσα κατάσταση. Συγκεκριμένα με το Συγκεκριμένο ερώτημα που κάνετε σχετικά με την ε, ε, αστική ευθύνη. Ε, οι κανονισμοί δεν αφορούν συγκεκριμένες εταιρείε, αλλά ισχύουν για όλους τους σχετικούς οικονομικούς τομείς. Υπάρχουν εθνικά πρότυπα τα οποία πρέπει να επιβάλλουν τα κράτη-μέλη σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να στραφώ στις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες για να σας πω ότι και εγώ και η ομάδα μου, ε, η ομάδα μου Είμαστε ικανοποιημένοι που ακούμε για την πρόοδο που γίνεται για τη συμφωνία SWIFT με την οποία ασχοληθήκαμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπαρόζο να μας πει τι χρήσιμα διδάγματα άντλησε η Κομισιό από τη συμφωνία SWIFT που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επωφελώς όταν θα ασχοληθούμε με τις συμφωνίες PNR που θα μας απασχολήσουν με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες πρώτα και μετά με τον Καναδά και την Αυστραλία. Ίσως είναι πολύ νωρίς για να αντλήσουμε διδάγματα, διότι δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει την διαδικασία. Περιμένουμε να αποπερατωθεί όλη αυτή η διαδικασία με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι χωρίς αυτή την υποστήριξη δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι το θέμα της ασφάλειας σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων. Είμαστε προσιλωμένη σε αυτά και πιστεύουμε ότι η συμφωνία όσο έχει τώρα μπορεί να απαντήσει στις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει όμως ένα πιο γενικό σημείο το οποίο εσείς υπογραμμίσατε. Είναι η σημασία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι ο σημαντικότερος εταίρος ε, της Ευρώπης. Πολιτικά λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνάψουμε αυτήν την συμφωνία. Ο πρόεδρος Biden ήρθε εδώ ε, και υπερασπίστηκε ε, τις διατλαντικές σχέσεις ακόμα και στον τομέα αυτό. Η Κομοσιό δεν θα συνιστούσε μια θετική ψήφο αν δεν ήταν πεπισμένη ότι είναι προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών για τη δική μας ασφάλεια αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό ως σήμα ε, της δέσμευσής μας για τις καλές σχέσεις με τον μεγαλύτερο εταίρο μας. Πρόσθετη ερώτηση. Συμφωνώ πλήρως κύριε Πρόεδρε με αυτό νομίζω ότι η συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελευταίως κυρίως υπήρξαν καλή δημοκρατική συμπεριφορά, καλό παράδειγμα για όλους. Η συμπληρωματική ερώτηση ε, τώρα είναι ε, πώς μοιράζεται ο φόρτος της εργασίας, η ευθύνη σχετικά με την τρομοκρατία ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συμφωνίες που συζητούμε μήπως επιβαρύνουν πολύ τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, σε σχέση με εμά με τον φόρτο που εμείς θα αναλάβουμε και τις ευθύνες και τους πόρους που θα διαθέσουμε για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Είναι σημαντικό αυτό το ε, σημείο. Οι Αμερικανοί μας είπαν ότι είναι έτοιμοι ε, να μας υποστηρίξουν αν θέλουμε να έχουμε ένα παρόμοιο σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η απόφαση που πρέπει να λάβουμε εδώ ε, στην Ευρώπη. Εμείς δεχόμαστε να παρέχουμε ε, δεδομένα, στοιχεία και υποστήριξη στις Αμερικανικές αρχές. Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στο σύστημα μας εμείς και οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι να μας βοηθήσουν τεχνικά διότι έχουν περισσότερες επενδύσεις στον τομέα αυτό από εμά και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε στο μέλλον διότι νομίζω όλοι μας πρέπει να ε, συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Δεν νομίζουμε ότι αυτή είναι αμερικανική ευθύνη και ότι εμείς την υποστηρίζουμε. Είναι κοινή ευθύνη να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και να προστατεύσουμε την ασφάλεια όλων των πολιτών μας. Η κυρία Γκαμπριέλε Τσίμερ παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα την έκθεση Κάσμαν ενέκρινε για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας για την ανάπτυξη. Ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εμάς είναι το ότι φυσικά θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε όλοι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκλίνουν ώστε οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη να μπορέσουν να επιτευχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν τήρησαν όμως τις υποχρεώσεις τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε έλλειμμα 20 δισεκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχουμε αναλάβει. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε εσείς κύριε Πρόεδρε, τι λαμβάνοντας υπόψη την σύνοδο του Συμβουλίου σκοπεύετε να κάνετε ώστε ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη να θυμηθούν αυτές τις υποχρεώσεις τους. Τι θα γίνει για να αυξηθεί η πίεση ώστε στην διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια ενωμένη εικόνα και λόγω της κρίσης που υπάρχει στα κράτη-μέλη να μην αποκλίνουν τα κράτη-μέλη από τις υποχρεώσεις τους. Ένα μέγεθος, ένας αριθμός ενό δισεκατομμυρίου ανθρώπων είναι εκείνο το μέγεθο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ζουν στη φτώχεια και στην πείνα αυτοί οι άνθρωποι. Συμφωνώ απολύτω με τι ανησυχίε που εκφράζεται. Υπάρχει όντω αυτή τη στιγμή ένα κίνδυνο λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών σε κράτη-μέλη κάποιε δεσμεύσει να μην γίνουν σεβαστέ. Ε, πράγματι, η Κομισιόν πριν από λίγε μέρε είχε μια συνάντηση στην Αντίσα Βέμπα ε, με την Επιτροπή τη Αφρικανική Ένωση. Και ένα από τα θέματα που έθεσαν οι εταίροι μα στην Αφρική είναι ότι μερικέ φορέ έχουν την αίσθηση ότι δεν γίνονται σεβαστέ οι δεσμεύσει μα. Υπάρχει λοιπόν θέμα πολιτική ε, υπευθυνότητα και από τη μεριά μα. Σίγουρα η Κομισιόν υποστηρίζει ε, να τηρήσουμε τι υποσχέσει μα ε, θα πάω στη Νέα Υόρκη. Ε, από τον Πάκη Μουν έλαβα χθες μια επιστολή ε, που υπογραμμίζει την σημασία αυτής της ατζέντα και θα το θέσω το θέμα όχι μόνο στην συνοδοκορυφή την ερχόμενη εβδομάδα αλλά και στους G20 και στον G8. Ο Γκλέν Ιγκλς είχα συμμετάσχει στη συνάντηση των G8 και εκεί επαναλήφθη η δέσμευση να κάνουν ό,τι έχουν υποσχεθεί. Ε, δεν έχω καμιά αμφιβολία βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν πάντα με ίδιες πρωτοβουλίε δραστηριοποιόταν ώστε να μπορέσει αυτό το έργο τη αναπτυξιακή πολιτική να το επιτελέσει. Για μένα όμως τίθεται το ερώτημα τι γίνεται σε σχέση με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, σήμερα, ώστε οι δομέ εκείνες, τα κονδύλια εκείνα, οι πόροι εκείνοι να, και οι προποθέσει να επιτευχθούν. Το, σημείο, το πρόγραμμα 12 σημείων που είχε συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Επίτροπο Πίμπαλξ να επιτελεστεί, να καλυφθεί. Τι κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεκτικότητα αυτών των πολιτικών. Για να δημιουργηθούν τα θεμέλια, να είναι συνεκτική αυτή η πολιτική. Και γιατί σε σχέση με αυτόν τον αγώνα, αυτή τη μάχη, αυτό δεν διαδραματίζει ρόλο στη στρατηγική 2020 από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν έχει αρμοδιότητα για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και πολλές φορές έχουμε ε, προτείνει στα κράτη-μέλη ε, προσθετή χρηματοδότηση. Ε, στην Ιαπωνία, παραδείγματος χάρη, του G80, ε, ε προτείναμε ένα δισεκατομμύριο επιπλέον χρηματοδότηση που θα μπορούσαν να προέρχουν και από τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια. Τώρα, για να τηρήσουμε τι δεσμεύσει μα ε, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα χρήματα πρέπει να έρθουν στο μεγαλύτερο ποσοστό από του εθνικού προπολογισμού. Με τι τρέχουσε δημοσιονομικέ προοπτικέ δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ευελιξία. Αυτό λοιπόν ε, κάνουμε, συζητάμε με τα κράτη-μέλη ώστε πραγματικά να τιμήσουμε τις δεσμεύσεις μας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω με ερώτηση για την ανάπτυξη και εν ώψη της Συνόδου του Συμβουλίου την Πέμπτη μεθαύριο. Η παρούσα οικονομική κρίση και η απειλούμενη ύφεση στην Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπιστεί κυρίως με αύξηση των επενδύσεων Βασικό μέλημα λοιπόν η εξασφάλιση πόρων χρηματοδότησης. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σκέφτεστε ως ε, πολιτικός ηγέτης της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης η Επιτροπή. Μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση έκδοσης ευρωπαϊκών ομολόγων για τη χρηματοδότηση μέγα ευρωπαϊκών αναπτυξιακών επενδύσεων Παραδείγματο χάρη, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, διευρωπαϊκή αυτοκινητόδρομη υψηλή ταχύτητα, διευρωπαϊκή έρευνα για τι κλιματικέ αλλαγέ, το e-health, πανευρωπαϊκό σύστημα ναυσιπλοεία ή μεγάλες επενδύσεις στην ενέργεια παραδείγματο χάρη LNG terminals στην Ευρωμεσόγειο. Μεγάλα ευρωπαϊκά πανευρωπαϊκού χαρακτήρα επενδυτικά έργα με έκδοση ομολόγων για την κάλυψή του. Uh, αυτά τα θέματα ελπίζουμε Ελπίζουμε ότι τα θέματα αυτά θα καλυφθούν από τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Για το 2020 έχουμε προτεραιότητες ό,τι έχουν σχέση με αυτές τις διασυνδέσεις, τις ενεργειακές, ε, των μεταφορών, ε, και τις ε, μορφές άειλης ε, διασύνδεσης όπως είναι η ατζέντα η ψηφιακή. Είναι οι τομείς οι οποίοι πιστεύουμε ότι θα έχουν προστιθέμενη αξία. Όπου ένα ευρώ που ξοδεύεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από ό,τι αν ξοδευτεί σε εθνικό επίπεδο. Διότι υπάρχει ένα συλλογισμό πίσω από αυτές τις επενδύσεις και από αυτή τη χρηματοδότηση. Πώς θα γίνει αυτό, αυτό πρέπει να συζητηθεί με τα κράτη-μέλη. Είναι δύσκολη εποχή τώρα να συζητήσουμε τους προϋπολογισμούς με τα κράτη-μέλη. Ε, μπορούμε βεβαίως να ζητήσουμε μεγαλύτερη διασύνδεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσθετη ερώτηση. Ότι δεν πήρα την απάντησή μου, δηλαδή πιστεύετε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο της ύφεσης με πανευρωπαϊκά συντονισμένες και άμεσες ενέργειες εκδίδοντας ευρωπαϊκά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά, η Ινδία, η Κίνα, η Αμερική, η Ευρώπη θα ανταποκριθεί με πανευρωπαϊκά μεγάλα, μεγάλες επενδύσεις. Θα παίξουν τα ευρωομόλογα καλύπτοντας αυτές τις επενδύσεις κάποιο ρόλο. Τι μπορεί να έχετε κατά νου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι τώρα υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουν τα κράτη-μέλη ευρωομόλογα για αυτά τα θέματα. Πρόσφατα ε, υιοθετήσαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, ένα μηχανισμό διευκόλυνσης για να βοηθήσουμε χώρες που έχουν προβλήματα χρέους είναι όντως ένα είδος, αν θέλετε, ε, υποχρέωσης ομολόγου ε, στις ε, χρηματοοικονομικές αγορές. Είναι δύσκολο τώρα να έχουμε ευρωομόλογα για αυτού του είδους τα έργα. Ωστόσο, νομίζω ότι υπάρχουν ορισμένες δυνατότητες χρησιμοποίησης άλλων μηχανισμών. Στο πρόγραμμά μου μίλησα ε, για ορισμένες ε, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέου για το πώς θα μπορούσε να συμμετέχει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εξετάζουμε όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης για αυτά τα πολύ σημαντικά έργα αλλά θέλετε την ειλικρινή ε, θέση μου. Είναι δύσκολο τώρα για να μην πω αδύνατο να έχουμε ευρωομόλογα για αυτά τα θέματα. Uh, Κύριε Πρόεδρε, Μπαρόσο, υποστηρίξατε την Βόρεια Ιρλανδία και τη σημαντική πρόοδο που επιτελέστηκε για να δημιουργηθεί ένα σταθερό μέλλον για το λαό μας. Στην έκθεση της Task Force υποδείξατε ότι υπάρχει υποστήριξη από την Κομισιόν για την δίκηση, την αποκεντρωμένη, την εξουσιοδοτημένη για ένα ευήμερο μέλλον για το λαό της Βορείου Ιρλανδίας. Σε αυτήν την εποχή η οικονομικής καχυξίας Νομίζω ότι υπάρχουν τομείς της οικονομίας στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι πάρα πολύ σημαντικοί, που υποφέρουν ε, από τις κυρώσει ε, για ε, ορισμένες παραβιάσεις που έχουν διαπιστωθεί από τους ελεγκτές για ε, την, το Υπουργείο Γεωργίας ε, και τις ε, μεταφορές για παραβιάσεις στα θέματα επιδοτήσεων γεωργών κυρώσεις είναι δυσανάλογες σε σχέση με τους κινδύνους για το όλο πρόγραμμα και υπάρχει μια πρόταση 5% καταποκοπή εφόσον ληφθούν μέτρα αμέσως από το Υπουργείο και τα χρήματα έχουν ήδη ανακτηθεί σε σχέση με τις αρχικές διεκδικήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα σχόλια σχετικά με την υποστήριξη της Κομισιόν προς τη Βόρεια Ιρλανδία. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις εξελίξεις και υποστηρίζουμε τις εξελίξεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Η Κομισιόν έχει επενδύσει πολλά σε αυτή τη διαδικασία. Θυμούμε την επίσκεψή μου στη Βόρεια Ιρλανδία και θα εξακολουθήσουμε να το πράττουμε. Ξέρω πολύ καλά το θέμα που αναφέρατε σχετικά με τις επιδοτήσεις και τις πληρωμές στους αγρότες. Έχει ήδη τονιστεί η θέση μας στο θέμα αυτό. Αλλά η καθάριση των λογαριασμών είναι μια προσέγγιση που υπάρχει. Το κάθε κράτος μέλος ε, μπορεί ε, να απαντήσει. Υπάρχει ανεξαρτησία της διαδικασίας. Δεν έχουμε διακριτική ευχέρεια ως προς ε, την, την διαδικασία αυτή. Πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση απέναντι στα κράτη-μέλη και πρέπει να τηρούμε πλήρως τους κανονισμούς όσον αφορά την λογοδοσία. Είναι κάτι το πολύ κρίσιμο, το σημαντικό. Σήμερα είχα μια συνάντηση με ε, ε, το ελεγκτικό συνέδριο και ήθελα να σας πω ότι ενώ υποστηρίζουμε την Βόρεια Ιρλανδία πρέπει να σεβόμεθα τους ε, κανόνες σχετικά με την λογοδοσία. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Um, Ευχαριστώ. Μια συμπληρωματική ερώτηση σε σχέση με αυτό. Υπάρχει κάποια ανησυχία στη Βόρεια Ιρλανδία ότι το ποσοστό μείωσης ε, βασίζεται σε μικρό ρυθμό σποραδικών ελέγχων μόνο. Θα ήθελα παρακαλώ ο Πρόεδρος να μας διαβεβαιώσει ότι η Κομισιόν θα κάνει την σωστή αξιολόγηση των διαδικασιών που ισχύουν ούτω ώστε το σχήμα να ε, ε, διοικείται σωστά, να εφαρμόζεται σωστά. Βεβαίω μπορώ να σα δώσω όλε τι εγγύσει εκ μέρου τη Κομισιόν ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια σωστή ε, ε, διαχείριση. Φυσικά όμω αυτή η διαδικασία είναι μια ε, διοικητική διαδικασία που περιλαμβάνει διάφορα βήματα. Περιλαμβάνει και δικαίωμα υπεράσπιση εκ μέρου του κράτου μέλου και δικαίωμα διαμεσολάβηση από έναν εξάρτητο τρίτο. Σας ευχαριστούμε πολύ και ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και περνάμε τώρα σε ένα συγκεκριμένο θέμα θεματολογικά. Η Task Force, η ομάδα κρούσης για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διακυβέρνησης. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Ο συνάδελφος θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Η συνάδελφος, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε Μπαρόζο, εσείς ε, σαφέστατα είπατε ένα πράγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η οικονομική κυβέρνηση της Ευρώπης. Το αναφέρατε. Όμως, περισσότερη κοινοτική μέθοδο. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε όταν θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση. Είμαστε δίπλα σας, στο πλευρό σας. Όμως στο Συμβούλιο υπάρχουν και διαφορετικές άλλες απόψεις ώστε μια διακυβερνητική μέθοδος να υιοθετηθεί, λέγεται όταν πρόκειται για παράδειγμα για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αν δούμε αυτή την μονάδα κρούσης Task Force και τα αποτελέσματα. Τι πιστεύετε ότι είναι τα πιο σημαντικά συμπεράσματα, ποια είναι αυτά που θα πρέπει να υπάρχουν στα συμπεράσματα, ώστε να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση και να ενδυναμωθεί το, σύστημα σταθερο... το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης με μια κοινοτική μέθοδο, με την κοινοτική μέθοδο. Συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να αναφέρετε. Καλό θα ήταν για τη συζήτηση αυτό που διεξάγεται και στους πολίτες. Ε, Ευχαριστώ. Η ομάδα δράσης δημιουργήθηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υποστήριξης προς την Ελλάδα και όπως ξέρετε η Κομισιόν συμμετείχε με απολύτω επικοδομικό τρόπο σε αυτήν την ομάδα δράσης. Η ομάδα δράσης μάλιστα ε, δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε συνεργασία με την Κομισιόν. Η Κομισιόν λοιπόν συμμετέχει στην ε, Task Force, στην ομάδα δράσης και μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι που προχωρεί ε, στις εργασίες της η ομάδα δράσης. Αναφέρεται μια ε, μορφή συνένεσης σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον οικονομικό συντονισμό στην Ευρώπη και τα περισσότερα από αυτά τα βήματα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις προτάσεις που γίνονται στην ανακοίνωσή μας το 12 Μαΐου. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η ομάδα δράσης ε, αποδίδει σημαντικό έργο γιατί ασχολείται με σημαντικά θέματα όπως είναι η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και περιμένουμε με ανυπομονησία ε, την πέμπτη, την πρώτη έκθεση που θα γίνει προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Φυσικά η Κομισιόν έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας να, ε, και έχει το δικαίωμα να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις με βάση τη συνένεση που φαίνεται να δημιουργείται σε αυτήν την task force. Η κυρία Ελσβιέτα Ρουκατσέφκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Γνωρίζουμε για τις δυσκολίες, οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη και πώς αυτό επηρεάζει τα αισθήματα των πολιτών αυτών των χωρών και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Πρόσφατα ακούσαμε για την ανάγκη να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όσον αφορά τα 27 κράτη-μέλη. Σας ερωτώ όμω πώς θα υπερασπιστείτε αυτή τη θέση και πώς θα συνεργαστείτε ώστε να υπάρξει πίεση για την εισαγωγή και υιοθέτηση νέων ε, προτάσεων και λύσεων για μια οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης όταν στην Ευρωζώνη αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ποιε εγγυήσει, ποια εχέγγυα μπορείτε να δώσετε όσον αφορά χώρε που ε, καταβάλουν τέτοιε προσπάθειε υπέρ τη οικονομική ευρωστία του ότι δεν θα καταλήξουν στη δεύτερη κατηγορία χωρών. Πρώτα με ότι είμαστε εναντίον ε, παράλληλου ανταγωνισμού αποφάσεων που είναι παράλληλος ανταγωνισμός ε, των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με τα θεσμικά μας όργανα, με 27 κράτη-μέλη σήμερα και βεβαίως πρέπει να τηρούμε πλήρως ε, τις συνθήκες. Δεν μπορούμε με το παρόν πλαίσιο να κάνουμε περισσότερα για τον οικονομικό συντονισμό και έχουμε τη συνθήκη, το άρθρο 121, το οποίο σαφώς θεσπίζει ότι η οικονομική πολιτική των κρατών μελών είναι μέλημα ευρωπαϊκό, αλλά είναι έργο των κρατών, είναι έκκληση για συντονισμό. Έχουμε και το άρθρο 126 ε, το οποίο αναφέρεται στις δημοσιονομικές πολιτές και το 136 που επιτρέπει στην Κομισιόν να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ενισχύσει τον συντονισμό και στην Ευρωζώνη και γενικά στο πλαίσιο το κοινοτικό. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε προτάσεις για την Ευρωζώνη αλλά πάντοτε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι η Ευρωζώνη είναι κάτι το ξεχωριστό από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κρίσιμο και σημαντικό για την επιτυχία της Ένωσης που βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης. Ευχαριστώ. Ο Σέρτζο Κομφεράτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μία γνώμη διαφορετική κάπως από αυτή του Προέδρου Μπαρόζο σχετικά με τις εργασίες των τελευταίων μηνών στην Κομισιόν και στην Task Force. Έχω μία σαφή αίσθηση και θα ήθελα να με διαψεύσετε ότι ε, έχει υλοποιηθεί και με, από ό,τι φαίνεται και στα μίντια ε, η ιδέα Τη εξυγίανση των ε, δημοσιομικών των κρατών μελών. Πράγμα το οποίο υποστηρίζω βεβαίω, αλλά αντίθετα αποδυναμώθηκε πάρα πολύ η, ε, ιδέα τη ε, ανάπτυξης και της μεγέθυνσης. Δηλαδή το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης φαίνεται να μείνει μόνο σύμφωνο σταθερότητας αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Ε, πρέπει λοιπόν να αναλυφθούν δράσεις ξεκινώντας από τη δημιουργία ευρωομολόγων που θα προωθήσουν την ανάπτυξη. Ε, γιατί ε, θα πρέπει η, πραγματικά η ανάπτυξη να είναι ενδιαφέρον και της Task Force και της ίδιας της Κομισιόν. Η ομάδα δράσης ασχολήθηκε με την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό ήταν ο ρόλος της. Και μέχρι τώρα σε αυτό αναφέρθηκα. Βεβαίω η ανάπτυξη είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Η ανάπτυξη είναι το πιο σημαντικό θέμα για την, ανα... για την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρί ανάπτυξη δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτά που περιμένουν οι πολίτε μα. Δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την ε, κοινωνική ε, ε, οικονομία τη αγορά. Δεν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πλήρω το δυναμικό μα. Αυτό ακριβώ είναι και το 2020. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και ανάπτυξη. Όχι όμως οποιαδήποτε ανάπτυξη, ε, ανάπτυξη, αϊφόρος ανάπτυξη ε, που θα περιλαμβάνει τους πάντες. Βεβαίω για την ανάπτυξη χρειάζεται εμπιστοσύνη. Και χωρίς να επανέλθει η εμπιστοσύνη στις, δημοσιομικές, στις τη αγορές Ένωση, Ευρωπαϊκής δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικά τα δημοσιονομικά και φορολογικά μέσα. Όχι σαν αυτός σκοπός, αλλά σαν μέσο για να επιτύχουμε μεγαλύτερα ε, επίπεδα ανάπτυξη για να αυξήσουμε το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Συνάδελφο Σιέτ Καμάλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη υγιούς οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που είδαμε είναι κατάφορη παραβίαση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, και έχουμε διάφορες δραστηριότητες και μοντάζ χρηματοοικονομικά δραστηριότητες έξω δημοσιονομικές. Χρειαζόμαστε υγιείς πολιτικές ε, λογοδοσία ε, λογιστικά πρότυπα. Αλλά αυτό μήπως ε, θα αντιμετωπίσετε το πραγματικό πρόβλημα των χωρών ε, που έχουν μεγάλο χρέος αντί να εστιαστείτε στην αύξηση της εξουσίας σας απάνω στους προπολογισμούς των κρατών μελών. Δεν το βλέπω το θέμα από αυτήν την άποψη. Δεν είναι ένας αγώνας για περισσότερη εξουσία. Όχι, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό που έχουμε τώρα και έχουμε το άρθρο της συνθήκης που είναι σαφέσα, ήδη τώρα η οικονομική πολιτική των κρατών μελών δεν είναι μόνο θέμα ε, εθνικού, ε, εθνικής επιδίωξης και μελήματες. Είδαμε ότι αυτό που συμβαίνει σε μια χώρα έχει σημαντικές επιπτώσεις πάνω στις άλλες χώρες. Έχει λοιπόν νόημα τα κράτη-μέλη όταν προετοιμάζουν τους προϋπολογισμούς τους να ξέρουν τι κάνουν οι άλλοι, διότι οι συνέπειες των αποφάσεων ενός κράτους έχουν, ε, έχουν συνέπειες πάνω στα άλλα κράτη. Δεν θέλουμε εμείς να παρεμβαίνουμε στα κυριαρχικά δικαιώματα και αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων. Πρέπει να σεβόμαστε τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά νομίζω ότι όταν συζητούμε την οικονομική πολιτική για την Ευρώπη, βλέπουμε πόση αλληλεξάρτηση υπάρχει, να ξέρουμε ποιες είναι οι προθέσεις των διαφόρων οικονομιών. Και αυτό είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία του να είμαστε μαζί και γι' αυτό η Κομισιό προτείνει κάτι και νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κονσένσους σύμφωνα με το πνεύμα αυτό. Κυρία Ενίκο Γκιούλη. Ναι, θα θέλουμε να δείξουμε ότι η Ένωση δεν έχει χρόνο να χάσει. Πρέπει να αντιδράσουμε αμέσως. Υπάρχουν τρεις τομείς όπου πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα. Η διακυβέρνηση, η στρατηγική της ανάπτυξης και η μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν χωρίς να ξεχνούμε ότι η πολιτική συνοχή, η αγροτική πολιτική που έχουν ε, καλά αποτελέσματα πρέπει να έχουν τη θέση τους. Χωρίς συνοχή και χωρίς ε, τα διατροφικά προϊόντα δεν μπορούμε να είμαστε ισχυροί στον κόσμο. Ζητώ από τον πρόεδρο της Επιτροπής. Ε, έχετε δεσμευθεί στην, για την στρατηγική 2020 να είναι εναρμονισμένη με αυτές τις πολιτικές και ως υπεύθυνο θέλετε να διατηρήσετε στους τρεις τομείς στην αρχή ότι όλες οι αλλαγές δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν παρά μόνο με αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο ε, τις χώρες της Ευρωζώνης χωρίς να φύγεται η συνοχή. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν ε, αναφέρεστε σε μια ολιστική προσέγγιση. Υπάρχουν λάθη και νομίζω ότι οι χώρε μέλη το έχουν συνειδητοποιήσει. Αυτό όταν μιλάμε για την οικονομική πολιτική στην Ευρώπη, όταν μιλάμε για το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, είναι μόνο ένα θέμα αυτό. Ε, θέλουμε να έχουμε οικονομική μεγέθυνση. Για να έχουμε εφορία πρέπει να έχουμε υγιή οικονομική διακυβέρνηση, να σεβόμαστε το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, να χρειαζόμαστε και νέου κανονισμού για τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ και πρέπει να επενδύσουμε στι δυνατότητε που έχουμε για ανάπτυξη. Για περί αυτού πρόκειται. Μεταρρυθμίσει, γι' αυτό επιμένω, χρειαζόμαστε δημοσιονομική εξυγίανση, σταθεροποίηση και πρέπει να συνεχίσουμε τι οικονομικέ πολιτικέ που είναι τόσο σημαντικέ για μα στην Ευρώπη από την άποψη οικονομική και κοινωνικής συνοχή. όχι για τους, μόνο τους 16 και τους 17, διότι, ε, αλλά για όλα τα 27 κράτη-μέλη. Ο κύριος παρακαλώ. με αυτή την ομάδα δράσης ο πρόεδρος Φαν Ρόμποϊ θέλει να επιταχύνει ώστε να μπορέσει η ευρώ να ε, εξέλθει από αυτή την οικονομική κρίση. Λοιπόν κύριε πρόεδρε επανειλημμένα σήμερα αναφερθήκατε στο άρθρο 121. Πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει αμοιβαία αλληλεξάρτηση και ότι φυσικά δεν πρόκειται εδώ για κάποιο ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο. Τώρα, σα ερωτώ συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό μέσα στην ίδια ομάδα δράση εξετάζεται η πιθανότητα επιβολή κυρώσεων έναντι κρατών που επανειλημμένα έχουν παραβιάσει αυτού του κανόνε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί σε σχέση με τι επιχορηγήσει και ή τα μέτρα ενίσχυση στα διαρθρωτικά να ε, ε, επιβάλλει κάποιε κυρώσει. Τι θα είχατε υπόψη σα ε, και ποιε δυνατότητε υπάρχουν για την επιβολή αυτών των κυρώσεων και πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ενιαία ρύθμιση για κράτη τα οποία δεν είναι ικανά πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ. Θέσετε πολλά ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που κάνουμε τώρα στην ομάδα δράσης και η ίδια η ανακοίνωση της Κομισιόν της 12ης Μαΐου το ανέφερε αυτό. Μιλάμε για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και με την διεύρυνση του οπλοστασίου που έχουμε ε, με κίνητρα για συμμόρφωση. Έτσι τα ονομάζω εγώ. Κάποιοι μιλάνε για κυρώσει βέβαια, εμεί μιλάμε για κίνητρα συμμόρφωση. Χρειαζόμαστε όμω αυτά τα μέσα που θα επιβάλλουν το σεβασμό του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν ε, σέβονται τη συνθήκη που τα ίδια υπέγραψαν και επικύρωσαν. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε με δίκαιο τρόπο. Όχι ε, τιμωρώντα τι χώρε που είναι στο Ταμείο Συνοχή και γι' αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά τα κίνητρα συμμόρφωση ανεξάρτητα από το αν είναι κράτη συνοχή ή όχι τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Τώρα, για την επιβολή αυτών των ε, κινήτρων ε, συμμόρφωσης μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Παραδείγματο χάρη μπορούμε να τα ε, χρησιμοποιήσουμε σε μια προληπτική φάση, σε φάση πρόληψης, αλλά με ένα αυξημένο βαθμό αυτοματισμού. Και η Κομισιόν θα κάνει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Γουέν Λόπες Ακουίδο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Μπαρόζο, θα ήθελα να σας ακούσω να κάνετε λόγο για την ανεργία, για τους ανέργους όταν εξειδικεύετε τους στόχους ε, της ομάδας δράσης ε, για την οικονομική διακυβέρνηση. Διότι αναφερθήκατε επανειλημμένα στη στρατηγική για μια ευφυή ανάπτυξη και αηφόρο ανάπτυξη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη και πρέπει να είναι αηφόρος και ολοκληρωμένη. Έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων που έχουν εξωθηθεί εκτός εργασίας ε, σαν συνέπεια αυτή της ε, ομής κρίσης. Έχουμε εκατομμύρια ανέργων που θέλουν εξειδικευμένα μέτρα όταν αναφέρεται ότι η οικονομική λέει, διακυβέρνηση, η σταθερότητα και η εποπτεία, η επιτήρηση του πακέτου μέτρων θα αντανακλούν μια στρατηγική που θα στοχεύει άμεσα στο να επανενταχθούν στην εργασία αυτοί οι άνθρωποι με έναν ορίζοντα χρονορίζοντα μεγαλύτερης παραγωγικότητας και μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη. Σε όλα αυτά τα άτομα που πρέπει να ενταχθούν και που έχουν οι ίδιοι υποστεί τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης και ιδιαίτερα πώς θα αντανακλάτε στη συμμετοχή των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συμμετάσχουν σε αυτή την ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε και πώς θα καθοριστούν νέοι κανόνες για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση στην λέσχη των 20 που θα συνέρθει. Ευχαριστώ. Είναι θεμελιώδε αυτό το οποίο είπε ο Ευρωβουλευτή κ. Ε, Λόπεθ Αγγιλάρ. Πρέπει να έχουμε μια ολιστική σφαιρική προσέγγιση. Δεν μπορούμε να ε, κατακαιρματιζόμαστε σε επιμέρου θέματα. Πρέπει να δούμε το σύνολο εκείνου που μπορούμε να κάνουμε υπέρ τη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Κυρίω ε, για την ανάπτυξη τη αηφόρου πολιτική ανάπτυξη ανάπτυξη. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Θέλουμε το κόστο αυτή τη προσαρμογή ε, να μπορούν ε, οι πιο αδύναμοι να το επομισθούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να δούμε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει καλύτερη ανακατανομή αυτών των ε, βαρών. Και γνωρίζουμε, όπω είπε και ο κύριο Λόπεθ Αγγιλάρ, ότι είναι αναγκαίο να έχουμε μια εξωτερική διάσταση στι δράσει μα. Γι' αυτό θα πάμε στη λέσχη των 20, G20. Θα προτείνουμε ίσω εκεί κιόλα μηχανισμού για τη συνεισφορά του οικονομικού τομέα για αυτή την κρίση, προσπαθώντας να ενισχύσουμε και να βρούμε μια κοινή θέση της Ευρώπης στο παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτρου Λούχαν Σχετικά με την Ευρώπη 2020 είναι μια νέα στρατηγική για την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση μεταξύ των βασικών στόχων που εγκρίθηκαν το Μάρτιο στις 25 και 26 Μαρτίου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπάρχει και ο στόχος της βελτίωσης της έρευνας και της ανάπτυξης, ούτως ώστε οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα αυτό να φτάσουν στο 30% του ΑΕΠ και στην ίδια απόφαση λέχθηκε ότι η Κομισιό θα εκπονήσει έναν δίκτυ το οποίο θα αντανακλά ε, το ύψος της έρευνας και ανάπτυξη. Σύμφωνα με ποια μεθοδολογία θα εκπονήσετε αυτόν τον δίκτυ και δεύτερον υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα διαβουλεύσεων Λοιπόν, ε, για το σκοπό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Έχουμε αναφέρει στο 3%, 3 όχι 30, αλλά δεν έχουμε αναφέρει την έρευνα και ανάπτυξη, αλλά την αντίληψη της καινοτομίας, διότι δεν πρόκειται μόνο για την βασική έρευνα, αλλά για το πώς η έρευνα μεταφράζεται σε οικονομική δραστηριότητα. Τι μπορεί να κάνει η έρευνα για περισσότερη ανάπτυξη, για περισσότερη απασχόληση. Και όπως ξέρετε, δεν υπάρχει ένας δείκτης καθορισμένος για την καινοτομία. Είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο διχάζει τους εμπειρογνώμενες συζητήθηκε το θέμα αυτό στον ΩΣΑ και πάρα πολλοί εμπειρογνώμενε ήρθαν στις Βρυξέλλες πρόσφατα και συνεργαζόμαστε μαζί τους και με άλλους για να έχουμε ένα δίκτυ της καινοτομία που θα μπορούσε να συμφωνηθεί από την, ε, την ε, κοινότητα των επιχειρηματιών ε, και άλλων. Και θέλουμε αυτό να γίνει με ανοιχτές διαβουλεύσεις και χαιρετίζουμε όλες τις συμβολές και συνεισφορές για να έχουμε καλύτερους δείκτες για την καινοτομία. Η κυρία Ρίντα Φιγκερέντο. Σα ευχαριστώ. Είναι ανησυχητική αυτή η κατάσταση όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ ευάλωτη και είναι ανεπαρκής για να μειωθεί η ανεργία και να δημιουργηθεί απασχόληση όπως την χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές λιτότητας και οι τεράστιες υποχρεώσεις για την υλοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και των Κριτηρίων έχουν την αντίθετη κατεύθυνση από την ανάγκη της δημιουργίας απασχόλησης. Ε, επιδεινώνονται οι ανισότητες και η φτώχεια είναι εκείνη η οποία ε, διευρύνεται. Και γι' αυτό όταν βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της ίδιας της φτώχειας, εμείς τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι κατάσταση αποκλεισμού, κατάσταση φτώχειας, ε, προβλημάτων για το, τους πολίτες. Σας ερωτώ Πρόεδρε, δεν είναι κατεπήγον να δοθεί προτεραιότητα προτεραιότητα σε αυτές τις μακροοικονομικές πολιτικές ε, στην αηφορία των κοινωνικών μέτρων αντί να συνεχίσουμε να εμένουμε και να επιμένουμε στην οικονομική αηφορία που βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει αντίθετη κατεύθυνση από την κοινωνική αηφορία. Δεν πρέπει να αναθεωρήσετε αυτά τα κριτήρια τα οποία είναι παράλογο και να δοθεί προτεραιότητα στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Ευχαριστώ. Sem sustentabilidade financeira não teremos sustentabilidade social. Χωρίς ε, οικονομική βιωσιμότητα δεν έχουμε κοινωνική βιωσιμότητα. Γιατί χωρίς την οικονομική βιωσιμότητα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχουν επενδύσεις, χωρίς επενδύσεις απασχόληση. Οι σταθερές και υγιείς οικονομικές, ε, ε, μακροοικονομικές πολιτικές βοηθούν τη φτώχεια. Και ένα από του στόχου τη ε, στρατηγικής του Ευρώπη 2020 είναι η καταπολέμηση τη φτώχεια, ε, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, με αριθμητικού στόχου μάλιστα πολλέ φορέ. Νομίζω ότι σήμερα ο κίνδυνο αύξηση τη φτώχεια είναι μεγαλύτερο ακόμα. Έχουμε καινούργια φαινόμενα φτώχεια. Εξαιρετικά ανησυχητικά. Οπότε οι κυβερνήσει στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων του θα πρέπει να δουν η κάθε μία πώ θα απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα. Όμω η λύση επαναλαμβάνω, δεν είναι η δημοσιονομική απειθαρχία. Διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε χειροτέρευση της κατάστασης και μάλιστα των πιο φτωχών. Και ο Τζον Μπάφτον. <coughs> Uh, Κύριε Πρόεδρε Μπαρούσο, θα μπορούσατε να μου πείτε ποιος επωφελείται από το πακέτο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, ο ελληνικός λαός, ε, ή οι τραπεζίτες τύπου Σπυρουλάτσι που είναι ε, ο ιδιοκτήτης της τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας στην ε, Ελλάδα. Μήπως εκεί υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Ευχαριστώ. The package put forward. Το πακέτο ε, ωφελεί τον ελληνικό λαό και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα είχε εγκριθεί το πακέτο αυτό από τα 27 κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά ε, το υπονοούμενο, ε, δεν νομίζω ότι αξίζει απάντηση. Τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση συνενούν στο ότι η ευρωπαϊκή ένωση δεν έχει ανάγκη νέων θεσμών. αυτό τουλάχιστον φάνηκε από τι δηλώσει τη κυρία μέρκελ και του κυρίου σαρκοζή την περασμένη εβδομάδα. ωστόσο διαφαίνεται αναφέρθηκε και πριν πω οδεύουμε σε μια νέα τροποποίηση του συμφώνου σταθερότητα όπου θα επιβάλλονται κυρώσει όπω η άρση του δικαιώματο ψήφου σε κράτη μέλη που δεν τηρούν την πειθαρχία στο δημοσιονομικό πεδίο. η ερώτησή μου είναι απλή πιστεύετε ότι το πρόβλημα διακυβέρνησης της ευρώπης αντιμετωπίζεται και περιορίζεται σε θέματα πειθαρχίας σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική προσαρμογή ή τελικά εν μέσω κρίσης έχοντας το νομισματικό εργαλείο σε κοινοτικό επίπεδο και το δημοσιονομικό σε εθνικό καταλήγουμε σε αδιέξοδο. Έχουμε προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένως. Χθες μόλις ο οίκος Moody's για μια ακόμη φορά ανετιολόγητα υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος η διεύρυνση οπλοστασίου που μας είπατε θα μας οδηγήσει σε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν κάτι το αξιόπιστο για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξη. Είναι προφανές ότι υπάρχουν θέματα εφαρμογής, υλοποίησης, η μη τήρηση από κράτη-μέλη ορισμένων κανόνων που έχουν συμφωνήσει ε, ήδη τώρα με τις συνθήκες που υπάρχουν και χωρίς νέες μεταρρυθμίσεις μπορούν να υπάρξουν ορισμένοι περιορισμοί και ορισμένες κυρώσεις. Αυτό είναι δυνατόν, είναι εφικτό. Αυτό που θέλουμε στο μέλλον είναι να υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του συμφώνου αλλά με δίκαιο τρόπο. Τα μέτρα να εφαρμόζονται με αντικειμενικό τρόπο και ε, σεβόμενοι την κατάσταση της ε, κάθε χώρας είτε πρόκειται για χώρα πλούσια είτε για χώρα πτωχή. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να έχουμε έναν πιο αξιόπιστο τρόπο ε, υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ώρα αυτή των ερωτήσεων. Θα ε, συναντηθούμε και πάλι τον επόμενο μήνα την ώρα των ερωτήσεων και στις συζητήσεις αύριο. Ευχαριστώ πολύ.